Βλέπω ότι η αίθουσα είναι σχεδόν γεμάτη και αρχίζουμε με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Έχτες. Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το σημείο 15. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον θα πρέπει να το μεταθέσουμε για την επόμενη συνεδρίαση γιατί δεν έχουμε καιρό πια. Και προχωράμε στο σημείο 16, το πρωτεϊνικό έλλειμμα της ΕΕ. Πώς θα λυθεί ένα διαονιζόμενο πρόβλημα. Ε, διαδικαστικό πρόεδρε. Η χθεσινή συνάντηση πρόεδρε. Η χθεσινή συνάντηση που προεδρεύσατε εσείς ήταν πολύ ε, καλά οργανωμένη, πολύ επαγγελματική, αλλά για μια ακόμη φορά δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για τα θέματα της εφαρμογής. Δηλαδή, πολύ συχνά λέμε ότι ε, θα πρέπει οι νομοθετικές αποφάσεις να τίθενται σε εφαρμογή και πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την εφαρμογή τους και όταν τίθενται τέτοια θέματα τα βάζουμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης και για δεύτερη φορά δεν τα συζητάμε, δεν προλαβαίνουμε. Και φυσικά χάνεται ο χρόνος και ο δικός μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι η κατάσταση αυτή δεν σας αρέσει ούτε σε εσάς ε, μας είπαν ότι αυτά τα θέματα δεν θα τα συζητήσουμε ξανά παρά μόνο το Μάρτιο, θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες. Δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να βρείτε περισσότερο χρόνο συνεδρίασης και να μπορέσουμε τα θέματα αυτά να τα συζητήσουμε παρκώς. Συμφωνώ μαζί σας ίσως στους συντονιστές να τα συζητήσουμε γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ πρόβλημα χρόνου έντονο, έχουμε πολλούς υπουργούς που μας επισκέπτονται και δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ωράριο που έχει συμφωνηθεί μαζί τους. Αύριο το πρωί λοιπόν στους συντονιστές θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν στο 16 έλλειψη πρωτεϊνούχων. Ο Τσάμπα είναι ο εισηγητής μας. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 6, υπέρ. Τροπολογία 6. Κατά, άποχες, <clears throat> απορρίπτεται. Τροπολογία 5 με μια ε, διαχωρισμένη ψηφοφορία ε, υπέρ, το πρώτο μέρος, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Check. Check, Monsieur le Président, check. Mm. check Check m'allons check Checker, So, Abstimmung beendet. Ωραία. <clears throat> Τελείωσε η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η απορρίπτεται, ξεκάθαρα απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Επτά. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Εν συνεχεία έχουμε την τροπολογία C2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Από τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές. Ε. Ε, υπέρ 14. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η προηγούμενη εγκρίθηκε. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 17 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Ε, το C3 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Προχωράμε στην τροπολογία 25 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική C1 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 32 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, άποχες, Απορρίπτεται. Τροπολογία 1, στα εκτιμώντας, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Τροπολογία 2, εκτιμώντας, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 3, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 39 υπέρ ουδής κατά. 11 αποχές. Σερμά συγχαριστήρια στον κύριο Σάμπα για την γνωμοδότησή του. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης 17. Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Στρέλα, η συγγήτρια. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σύντομα, σύντομα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σύντομα, σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους σκιώδεις για τη συνεργασία που είχαμε που ήταν πολύ επικοδομητική και χρήσιμη και μας επέτρεψε να καταλήξουμε στους συμβιβασμούς που θα δείτε. Είχαν κατατεθεί 204 τροπολογίες από τις διάφορες επιτροπές και τώρα με, τους, με τις συμβιβαστικές μπορούμε να κάνουμε το κείμενο πιο συνοπτικό και πιο εύληπτο χωρίς επαναλήψεις. Δεύτερον, να σας πω μερικά σημαντικά για την ψηφοφορία, τουλάχιστον για την πορτογαλική μετάφραση που έχει ορισμένες ασάφειες στους τεχνικούς όρους και πρέπει να τους διορθώσουμε για να είναι το κείμενο και πάλι πιο εύληπτο. Εκεί που λέει εντατική περίθαλψη πρέπει να λέει διαφοροποιημένη περίθαλψη. Στο 198 ζητάμε ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι αυτό που γράφει εδώ. Α, ευχαριστούμε γλωσσικά λοιπόν θέματα είναι αυτά. Ναι, λέει ο πρόεδρος, η γλωσσολόγοι, εμπειρογνώμονες λύνουν τα προβλήματα αυτά τα γλωσσολογικά, τα μεταφραστικά. 72 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, <clears throat> απορρίπτεται, 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 24 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται, 75 υπέρ, κατά, Αποχές δεκτή. Επιτροπή ε, για γυναικείων υποθέσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 για την παράγραφο 2. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Ε, Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Προχωρούμε. Συμβιβαστική 4. 4 συμβιβαστική υπέρ. Κατά, άποχες, δεκτή. Προχωρούμε ε, με την ε, τροπολογία 18 υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές, δεκτή. 17 την Επιτροπή του Δικαιωμάτων των Γυναικών, κατά, αποχές, δεκτή. 89, 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 3β ΙΜΚΟ <clears throat> υπέρ κατά άποχες δεκτή ΙΜΚΟ 08 υπέρ κατά άποχες δεκτή ΙΜΚΟ 09 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Έχουμε μία τροπολογία consolidated, 6, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4b, 103. 103 τροπολογία, παράγραφος 4 νέα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 4β, ε, τροπολογία 103. Ήμκο 24. Δεκτή. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 106. 106. Abstimmung beendet. Πέρασε Ναι, χρειαζότανε. 28 υπέρ, 27 κατά. Δεκτή. 107 mm. υπέρ. Κατά. Α, δεκτή. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Ε, επόμενη σελίδα. 29 ε, Επιτροπή Γυναικείων Υποθέσεων. Ε, μη 29 υπέρ, κατά, δεκτή. 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ 157 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 120 και 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 122 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 129. Ε, να ελέγξουμε παρακαλώ. Α, το 122, συγγνώμη. 122 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή, δεκτή, 122. 129. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Ε, ε, ε, παρέμβαση, συγγνώμη, Εσείς ανακοινώσατε την 122 ενώ πρόκειται για την 129. Ναι, εμείς αυτήν ψηφίσαμε, γι' αυτό είχαμε μιλήσει. Ενώ εσείς ανακοινώσατε την άλλο άρθρο, όχι το ίδιο που είχαμε πει. Ε, κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στην ψήφιση του 122. Α, επαλήθευση για το 122 λοιπόν είχε ζητήσει η κυρία Ντεμπρόν, γι' αυτό το ζήτησα. Ναι, αλλά προηγουμένως μιλήσατε για την 129 και εμείς για αυτό ψηφίσαμε υπέρ. Ενώ επρόκειτο για το 122. Ναι, ε, εάν έγινε παρανόηση 122. Να ξαναεπαναλάβουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία 122 παρακαλώ. 122. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική. 122. Abstimmung ist beendet. Πέραση ψηφοφορία. Ναι, έγινε το μπέρδεμα, το, το δέχομαι λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε απορριφθεί, οπότε επιβεβαιώνεται. Τώρα είμαστε στην 129 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 132 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Επιτροπή γυναικών 105 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή η ε, Επιτροπή Γυναικών 14 η, κατά άποχες, δεκτή. 26 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 28 ε, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Θέλετε την 28. Ε, 28 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έληξε. Ε, έγινε δεκτή. Καθαρή πλειοψηφία. συμβαστική 11. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 143. 143. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 144. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Φαμ... Α, να ελέγξουμε την 144 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. Για 144. Παμ 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Φαμ 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήμκο 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήμκο 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήμκο 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήμκο 22 υπέρ κατά άποχες δεκτή Ήμκο 26 υπέρ κατά άποχες δεκτή Ήμκο 29 υπέρ άποχες δεκτή 151 υπέρ Άποχες. Απορρίπτεται. 152. Ε, υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 153. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 153. Έληξε πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπέρ. 155 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτεί. 160. Θέλετε να ελέγξουμε την 155 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία, δεκτή. 160 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Ήμκο 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ,

Α, καταπίπτει. Επειδή πέρασε η 163, άρα καταπίπτει. 165, Αντωνέσκου υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 166 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. ΦΑΜ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά άποχες δεκτή 130, 173 υπέρ κατά άποχες δεκτή 174 ε, υπέρ κατά Αποχές. Δεκτή. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 30 υπέρ κατά Α, Ξανά, ΦΑΜ 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ΙΜΚΟ 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή 184 υπέρ αποχές δεκτή 185 υπέρ κατά αποχές δεκτή 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή 188 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ε, 189 είναι γλωσσική διόρθωση. 190 υπέρ κατά άποχες. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 196 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 198 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 199 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 28 υπέρ κατά Αποχές. Δεκτή. Η 200 καταπίπτει. Προχωρούμε 201 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 23 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. ΦΑΜ 24 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήμκο 30 υπέρ, κατά, δεκτή. Ήμκο 32 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Η, η ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στις σιτασιόν. Ε, η ε, τρία. Η δύο έγινε δεκτή, η τρία δεκτή, η τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 δεκ, υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 δεκτή δεκτή 7 δεκτή υπέρ αποχές δεκτή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 δεκτές όλες φαμ 1, c 1 γ υπέρ κατά αποχές δεκτή ΦΑΜ 6 γάμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 γάμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκτιμώντας 1. Ε, στο 8, τροπολογία 8, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκτιμώντας τροπολογία 8, δεκτή. 10, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15. Ε, α, 15. Κατά πίπτη 16 επίσης. Ε, προχωρούμε στη συμβαστική Α, προχωρούμε με την 21. 21, τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23, υπέρ, κατά, Συγγνώμη, ψηφίζουμε 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 24 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 25 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Φαμ. Δι. Υπέρ. Η δέλτα. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Και 30 είναι ταυτόσιμη. Ε, συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. δεκτή. Δεν τελειώνει λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, 35. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΦΑΜ ή F. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 38. Υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 40. Ε, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 42. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 43. Υπέρ, κατά άποχες δεκτή. Επόμενη σελίδα, 49, <clears throat> υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 50, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 51, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 42, 52 ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ G υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Φαμ κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, θα ελέγξουμε την τροπολογία κάπα. Φαμ κάπα. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Τώρα είναι εντάξει, εντάξει. Οπότε, 31 υπέρ, 27 κατά. Δεκτή η τοπολογία ΦΑΜ, λαμ, φαμ καπα. Προχωρούμε. ΦΑΜ λάμδα. Λάμδα, L. ΦΑΜ, ε, υπέρ. Κατά, Αποχές. Φιλελεύθεροι, δεν βλέπω, παρακαλώ το λάμδα ξανά ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 55, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε με την 60, νέο εκτιμώντας, 60 τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή και έτσι τελείωσε ο μαραθώνιος και προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν μία ψήφο παραπάνω. Μία πρέπει να, να φύγει. Ακόμα, μία παραπάνω, μία πλεονάζει. Μία ψήφος πλεονάζει. οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες. Ε, μία ψήφος παρακαλώ. Περισσεύει. Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία, 52 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά, 7 αποχές, θερμά συγχαρητήρια κυρία Εστρέλα και σε όλους τους συνεργάτε. Ένα σημαντικό θέμα και πολύ επίκαιρο. Το τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. So, Επόμενη ψηφοφορία, επίσης ένα σημαντικό θέμα, το 18 αξιολόγηση της γρήπης 2009-2010. Συγγείτε η κυρία Ριβαζή. Ψηφίζουμε. Συμβιβαζιστική 1 νη 1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά περίοδο 2009-2010 ή συγείται η κυρία Ριβαζή. Ψηφίζουμε. Συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε. Στην ίδια σελίδα κάτω-κάτω συμβιβαστική 14. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Α, συμβιβαστική 86. Υπέρ, όχι, όχι συμβαστική, τροπολογία 86. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Τροπολογία 87 με προφορική τροπολογία. Και ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές δεκτό το πρώτο μέρος. Δεύτερο μέρος πίστη. Τροπολογία 89 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ε, τροπολογία 2, consolidated, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική, α, τροπολογία 100, υπέρ, 100. Α, απεσύρθη από τους συντάκτες, αλλά την ενέκρινε η εισηγήτρια. Την ψηφίζουμε. Τροπολογία 100. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 5 consolidated. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ναι, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Είναι 110. ε, πέρας της απορρίπτεται τροπολογία 6 consolidated υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 117 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 118. Την εγκρίνει η συγγήτρια. υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία, ε, συμβαστική 7. Υπέρ κατά, άποχες, δεκτή. Συμβαστική 8, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Τροπολογία 128, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται το ε, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Consolidated 10 υπέρ Λοιπόν, ένα αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας βάσει του κανονισμού 147 το 1 τέταρτο των μελών, δηλαδή 16 μέλη πρέπει να την υποστηρίξουν, 16. Οπότε έχουμε ονομαστική, βάσει του κανονισμού. Εάν 16 το δέχονται, το υπερψηφίζουν. Ακριβώς 16 είμαστε λοιπόν, βάσει του κανόνα 195 παράγραφος 3. 16 μέλη, οπότε κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία σε αυτό το consolidated 10, σε αυτή την τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 41 κατά, 2 αποχές, απερίφθη. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή Consolidated 11. Ψηφίζουμε την άλλη εκδοχή. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 173. Υπέρ. Ε, 137 συγγνώμη, αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 137 εγκρίθηκε. Consolidated 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 150 σε δύο τμήματα με ε, προφορική τροπολογία. Πρώτο μέρος παρακαλώ υπέρ. Ε, πρώτο μέρος της 150 υπέρ κατά Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο μέρος καταπίπτει. 151 επίσης σε δύο τμήματα, σε δύο μέρη. Ε, πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό, το δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. 152 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 153 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. σύμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 180 όχι 82 ή 82 ή 82 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 83. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 156 υπέρ κατά δεκτή. 161 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Consolidated 15 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 172 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ε, στα citations τώρα, τις παύλες, ε, ένα στα citation, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δύο, τροπο, ε, δύο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέντε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Έξι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεκτή. Συνεβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Consolidated 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τρίτο υπέρ, κατά, αποχές, επίσης δεκτό. Τροπολογία 23. Σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 24. Προφορική, με προφορική και ε, σε δύο τμήματα. Υπέρ, πρώτο τμήμα, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα ε, καταπίπτει. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά, άποχες, δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 37, τροπολογία 37, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 38, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 ε, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 51 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 22 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 55 τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 56, 57, 58 είναι ταυτόσιμες, ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Consolidated 23 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 66 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 67. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, άποχες, Απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 69-70 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 72. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία για την ε, γρήπη των χείρων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. 58 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στην κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ψηφοφορία η οποία είναι αρκετά επίκαιρη. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι σε περίπτωση πανδημίας να υπάρξει καλύτερη διαχείριση, ανεξαρτησία αλλά και συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ένα στοιχείο είναι οι λεγόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη Γαλλία αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων και σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γι' αυτό είχα ζητήσει να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να επισημαίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Πάντως ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη γραμματεία φυσικά της Επιτροπής, λέει η συγγήτρια. Έχουμε ακόμα το ερώτημα της συναδέλφου Ντελβού. Πράγματι χαίρομαι που καταλήξαμε τελικά στη διαδικασία αυτή με ένα κείμενο το οποίο λαμβάνει υπόψη γενικά όλων τις διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει το θέμα βέβαια της σύγκρουσης συμφερόντων αλλά γενικά υπάρχει μια ισορροπία. Θέλω να ευχαριστήσω σας και όλη συγγήτρια όλους όσους πήραν μέρος στην προσπάθεια. Υπάρχει κι άλλο ένα κείμενο, η αιτιολογική έκθεση, η οποία έχει παραμείνει ως έχει. Σύμφωνα με το άρθρο λοιπόν 52 του κανονισμού και στα πλαίσια μιας λογικής συνοχής θα έλεγα, θα ήθελα η αιτιολογική έκθεση αυτή να εξελιχθεί λιγάκι έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κείμενο το οποίο όπως υιοθετήθηκε θα ψηφιστεί ελπίζω και στην Ολομέλεια. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ λογικό να μην υπάρχει μια ασυνέπεια μέσα στο κείμενο. Θα πρέπει η γραμματεία να το ε, εξετάσει αυτό και μπορείτε όλοι μετά να το διαβάσετε αν συμφωνεί, αν είναι συμβατό το κείμενο. Προχωρούμε στο σημείο 19. Uh, εδώ τον κατάλογο Βλέπετε τι ωραία που φαίνεται εδώ ο κατάλογος της, ψηφο, της ψηφοφορίας που έχω στα χέρια μου. Δεκαεννέα. Η μέτρηση της πρόοδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Άννα Ρόσμπαχ. Έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους όσους συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή. Ακούστηκαν πολλά και θετικά, αλλά δυστυχώς χθε και σήμερα συνέλεξα αρκετές επιπλέον συστάσεις από πλευρά συναδέλφων οι οποίοι εμένουν στις θέσεις τους, κάνουν πόλεμο χαρακομμάτων θα έλεγα Νομίζω ότι δεν είναι η φάση τώρα να συζητάμε ε, με ιδεολογήματα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στον κατάλογο αναμονής θα έλεγα των προσυζήτηση θεμάτων. Είναι απαραίτητο να το συζητήσουμε. Η έκθεση αυτή είναι μια πρώτη φάση για μια σειρά άλλων πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να οριμάσουν. Εφόσον συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο βήμα, ή μάλλον εάν δεν προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε τότε δεν χρειάζεται να ασχολούμεθα πλέον με το θέμα. Εγώ δεν λέω τώρα ψηφίστε υπέρ ή κατά, αλλά το να καταψηφίσει κανείς αυτή την πρόταση δεν είναι σωστό. Ελπίζω να βρεθεί μια συνενετική λύση. Πρόκειται ε, για ένα πρώτο βήμα θα έλεγα και μετά θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην πιο ικανοποιητική μέθοδο για να συζητήσουμε το θέμα. Ας κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια να υπερψηφιστεί παρακαλώ το κείμενο. Ναι, πολύ ωραία. Ακούσαμε την εισηγήτρια, θα δούμε τώρα πώς θέλουν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι. Θα αρχίσουμε αμέσως με την τροπολογία 17, Βιτόριο Πρόντι, υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Της ε, οίκων 9 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι ε, πέρασε, αλλά να σας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 9. Έληξε ψηφοφορία. Α, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Τροπολογία 20, υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Δεν είναι σαφές. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 21 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Αγγλία. Α, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Διακόπτει ο πρόεδρος ένα λεπτό. Ε, εντάξει. Λύθηκε. Λοιπόν, 26. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση. Απερίφθη. Απορρίπτεται. Λοιπόν, 28 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οίκον 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εμπλουά. Ε, απασχόληση 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παρακαλώ να ελέγξουμε την Τροπολογία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η 34. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Είκον 14. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38. Υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Ε, 39 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 40. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έμπλ 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Οίκον 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία οίκων 16. Έλλειψη ψηφοφορία. Ίσα ίσα. Δεκτή. 28 έναντι 27. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καραπίπτη. Η 50, 50. Ψηφίζουμε την 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 27. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οίκον 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οίκον 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρα 3 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρα 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρα 10 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έμπλ, 6, 7, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Απασχόληση 7, υπέρ, 8, κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεκάξι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 17 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτό. Οίκον 15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτό. Έμπλ 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτό. Η πατροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Ξανά παρακαλώ. 52 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ε, ηλεκτρονικά τώρα. Έληξε. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 50. Τι είναι. 55 ηλεκτρονικά παρακαλώ. 55 ηλεκτρονικά. Έληξε. τσίμα τσίμα, αλλά πέρασε. Δεκτή. Η 55. Προχωρούμε. Είτε 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέγγι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οίκον 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. απολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 57 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άμπλ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές Α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική ψηφοφορία την 63 παρακαλώ. Έληξε ψηφοφορία δεκτή. Εκπίπτει 65, καταπίπτει 65. Όχι. Α, ψηφίζουμε την 65 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ την 65. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ απλώ 1 ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 9. Ε, Άμπλ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκτή. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οίκον 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέτζι 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 3. Υπέρ. Κα... Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέτζι 4. Υπέρ. Κατά. Ε, ε, πάω πολύ γρήγορα λέει ο πρόεδρος. Την 4. Regional, τη 4, Regi 4, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Έληξα. Απορρίπτεται. Η 4. Ρέγγι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, ελέγχουμε την πέντε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Έληξε. Δεκτή. Ρέγγι έξι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Ρέγγι 7, υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 7. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 83 και η 9 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεκτές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ η τροπολογία 83 και η 9. Έληξε ψηφοφορία είναι σαφές. Δεκτές, δεκτές. Προχωρούμε. Ρέγγι 8. Όχι, Ρέγγι 9, συγγνώμη. Ναι. Υπέρ. Ρέγγι 9. Ρέγγι 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οίκον 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οίκον 12 καταπίπτει. ΔΕΒΕ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 4. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, άποχες, δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύε 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύε 6 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτό. Δεκτή. Οίκον 10. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Τσεκ λοιπόν. Ηλεκτρονικό. Ή 10. Οίκον 10. Έλ, έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. Οίκον 13 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Έμπλ 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήτρα 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήτρε 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 70 υπέρ, Α. Α, τσεκ την 68, ηλεκτρονικά την 68 λέει τώρα ο πρόεδρος. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή η 68, δεκτή. 70 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 71, υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά άποχες δεκτή 76 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ. 81 δεκτή λέει ο πρόεδρος. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ την 81. Έληξε. Απορρίπτεται και μάλιστα σαφέστατα. 82 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 84 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Για την 85. Έληξε. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα, εκτιμώντας και παύλες. Ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή Citation 2 Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Citation Παύλα 1 Έμπλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Citation 2 Έμπλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προχωρούμε στο εκτιμώντας α, τροπολογία 5, πρώτη, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7, υπέρ. Κατά, αποχές, Δεκτή. Θέλετε... Όχι, είναι σαφές. Ε, τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ α, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήτρε α, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή check. Αν θέλετε, λέει ο πρόεδρο, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 10, η 10. Έληξε. Δεκτή, δεκτή. Η τροπολογία 10. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. κατά αποχές. Να ελέγξουμε τη 14 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έληξε. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έμπλ Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ε, δεκάξι, Τροπολογία δεκάξι, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έμπλ Σ. Γάμα. Υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται η έμπλ C, ήτρε C γάμα. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ε, ε, έμπλ δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήτρε D, δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και τελειώσαμε την ψηφοφορία για αυτή την έκθεση και ψηφίζουμε την έκθεση. Την τελική ψηφοφορία τώρα παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Έληξε η ψηφοφορία. 15 υπέρ, 34 κατά, 11 αποχές. Άρα δυστυχώς στον κάλαθο των αχρήστων πάει η έξεση. Η κυρία Ρόσπαχ, συγγήτρια. Το είχα πει από την αρχή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ψηφίσουμε για να καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων η όλη προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος αναχωμάτων όπως έλεγα προηγουμένως. Προσπαθώ να είμαι πραγματίστρια, προσπαθώ να δω τι μπορεί να διασωθεί, τι μπορεί να σημαδέψει το άνοιγμα αυτό προς μια νέα πορεία. Μια πορεία η οποία να μην λαμβάνει υπόψη μόνο το ΑΕΠ. Πάντως η πλειοψηφία της Επιτροπής μας εξέφρασε την άποψή της, θα πρέπει να δοκιμάσουμε με διαφορετικό και πιο πιστικό τρόπο στο μέλλον. Η μάχη η οποία δόθηκε ήταν μάχη η οποία ήταν αυστηρά ιδεολογική και αυτό είναι λυπηρό. Ε, δυστυχώς η πολιτική δεν εγγυάται και επιτυχία. Ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω σαν σκιώδη εισηγητής της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας. Εγώ από τη θέση μου προσπάθησα να μπω στην ουσία του εγγράφου αυτού ακριβώς γιατί κατανοούσα τη μεγάλη σημασία. Είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο που θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις αλλαγές που έχουμε μπροστά μας και πώς τα όρια των φυσικών πόρων και η δυνατότητα της γης και του περιβάλλοντος να απορροφά τα δικά μας προϊόντα πρέπει να αλλάξει. Απαιτείται μια αλλαγή σκέψης, μια αλλαγή πολιτισμού. Υπάρχουν όρια στη φύση και τα όρια αυτά δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν αυστηρά από το ΑΕΠ. Γιατί αυτό καλύπτει μόνο την υλική παραγωγή. Απαιτείται λοιπόν μια πολιτισμική αλλαγή η οποία να λαμβάνει υπόψη τον καθορισμό των κοινών αγαθών, των άειλων κοινών αγαθών, που βοηθούν τον πολιτισμό μας να κάνει άλματα προς τα εμπρός, και που ταυτόχρονα μπορούν να συνεισφέρουν στην αηφορία της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε και να περάσουμε από τα αυστηρά τρέχοντα υλικά αγαθά και στην κατανάλωση κάποιων αγαθών τα οποία θα χαρακτήριζα άειλα Έπρεπε να το κατανοήσουμε, δεν έγινε κατανοητό αυτό, ελπίζω να γίνει στο μέλλον. Μάλιστα. Έχει ήδη έρθει ο προσκεκλημένος μας, αλλά έχει ζητήσει το λόγο πρώτα η κυρία Λεπάζα. Σύντομα όμως, ε, σύντομα, σύντομα. Ναι κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια και εγώ σκιώδης της ομάδας μου, των φιλελεύθερων δηλαδή, κατάλαβα ότι έχει γίνει μια προσπάθεια τορπιλισμού της έκθεσης αυτής ενώ το θέμα είναι πολύ σημαντικό και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Πρόντι. Σε αυτά τα θέματα πάντοτε το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε, δηλαδή η απόρριψη της έκθεσης αυτής μπορεί να ερμηνευτεί ως ότι το κοινοβούλιο μας δεν δίνει σημασία στο θέμα. Νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι τροπολογία την τροπολογία θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει σε συμβιβασμό αν αποτύχανε βέβαια η προσπάθεια τορπιλισμού που έκανε η Ρέγγι. Πολλές σωστές τροπολογίες εγκρίθηκαν, αν και δεν τις εγκρίνω όλες. Εγώ ήμουν πάντως υπέρ γενικά της έκθεσης και κατάλαβα ότι έπεσε στον κάλαθο των αχρήστων δεν ξέρω αν μήπως το κοινοβούλιο δεν πρέπει να ξαναθίξει το θέμα με άλλο τρόπο. Να μην παραμείνουμε μόνο στο ΑΕΠ για να ε, κρίνουμε τις προόδους της κοινωνίας μας. Είναι παράλογο. Μάλιστα. Ο κύριος Σνέλχαρτ. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σημαντικό το θέμα. Αυτό το δεχόμαστε όλοι. Αλλά για να κρίνουμε ένα σοβαρό θέμα πρέπει να έχουμε σοβαρά και μετρήσιμα κριτήρια. Δηλαδή κριτήρια όχι υποκειμενικά αλλά αντικειμενικά. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε, γιατί θέλουμε συγκεκριμένα στοιχεία, λιγότερη γραφειοκρατία και γιατί είμαστε υπέρ της αποτελεσματικότητος, πράγμα που δεν το επέτρεπε η έκθεση αυτή. Το ΕΛΚ θέλει πάλι να μιλήσει. Όχι για το ίδιο θέμα κύριε Πρόεδρε. Είναι σχεδόν 11 και σας ζητώ ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να κάνουμε μία μικρή εσωτερική διαβούλευση μετά από αυτή τη μαραθώνια ψηφοφορία να έχουμε πεντάλεπτο ή εξάλεπτο διάλειμμα ή 6,5 λεπτό μέχρι να έρθει ο Ούγγρος Υπουργό των Εθνικών Πόρων που θα μας μιλήσει για θέματα υγείας. Το θέμα του επίσης είναι πολύ σημαντικό. Α, το θέμα που μόλις χειριστήκαμε είναι σημαντικό. Δεν λύγει εδώ η υπόθεση, αλλά παρακαλώ να ξανάρθετε για να ακούσουμε και τις απόψεις της Προεδρίας για τα θέματα υγείας. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από το σύντομο διάλειμμα, μετά από αυτό το μαραθώνιο των ψηφοφοριών, ερχόμαστε τώρα στην ε, πολύ σημαντική συνεδρίαση του πρωινού και χαιρετίζω τον ε, Υπουργό εθνικών πόρων της Ουγγαρίας, τον κύριο Μίκλος Ρέτζελη και χαιρετίζω και τους ε, συνεργάτες του που είναι υπεύθυνοι ε, στον τομέα της υγείας. Ε, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, είμαστε υπεύθυνοι, εμείς ασχολούμαστε με θέματα περιβάλλοντος, αλλά δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων επίσης και θα θέλαμε, περιμένουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το πρόγραμμά σας ε, της, ε, του επόμενου εξαμήνου και μπαίνουμε κατευθείαν στην ουσία και σας δίνω το λόγο για την παρουσίαση του προγράμματος της Ουγγρικής Προεδρίας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι παρόν σήμερα ανάμεσά σας για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα για την υγεία της Ουγγρικής Προεδρίας. Χαίρομαι που θα μπορέσω να εκφραστώ γύρω από τις πρωτοβουλίες που είναι στην ημερήσια διάταξη στον τομέα της υγείας. Από τότε που η Ουγγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει αρκετές εξελίξεις τα τελευταία 5-6 χρόνια όχι μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν σημαντικότατες αλλαγές και στον τομέα της συνθήκης, μέσω δηλαδή της συνθήκης της Λισαβόνας, αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου θεμελιώνεται σε νέες βάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κοινέ λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα επί των οποίων θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις σημαντικές τους επόμενους μήνες. Όπως είπα, τις τελευταίες έξι χρόνους διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας κατέστησαν σημαντικές. Πάντα παραμένουν οι εθνικές αποφάσεις σημαντικές στον τομέα της υγείας, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία απαιτούν απάντηση από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ευθύνε οι οποίες ε, σαν παράδειγμα άπτονται της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει καλύτερη συνεργασία όχι μόνο γιατί οι δυσκολίες είναι κοινέ, αλλά γιατί δυστυχώς υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής της υγείας και γενικότερα της κατάστασης της υγείας των πληθυσμών. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, όπως είπαμε, το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα στις ε, ε, υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Η διατήρηση και η αποκατάσταση της υγείας των πολιτών επηρεάζει φυσικά άμεσα και απόλυτα την ποιότητα ζωής του πολίτη και της κοινωνίας. Η προστασία της υγείας λοιπόν είναι αναπόσπαστο κομμάτι ακόμα και της ίδιας της οικονομικής διαδικασίας. Η υγεία του πολίτη, η υγεία του εργαζομένου, η υγεία ιδιαίτερα των πολιτών μιας κάποιας ηλικίας επηρεάζουν έναν πολύ μεγάλο τομέα της οικονομίας μας. Ο τομέας της υγείας προσφέρεται στην καινοτομία, προσφέρεται στην έρευνα, ευνοεί και ευνοείται από την τεχνολογική ανάπτυξη και ταυτόχρονα ο τομέας της υγείας είναι σημαντικός πελάτης σε εισαγωγικά για προϊόντα του τομέα της τεχνολογίας. Επίσης ε, και ε, σε επίπεδο απασχόλησης 10% ε, γύρω από την, της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέση με την υγεία. Στα πλαίσια της στρατηγικής λοιπόν για το 2020, τις προοπτικές δηλαδή για το μέλλον, η οικονομική ανάπτυξη καλείται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η υγεία του ενεργού πληθυσμού είναι ε, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και εδώ οι ευθύνε μας είναι και αυτές σημαντικές. Η Ουγγρική Προεδρία έρχεται σε μια δύσκολη οικονομικά στιγμή στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική κρίση έχει καταστήσει τις προκλήσεις ε, πιο δύσκολες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε φαινόμενα όπως η γύρανση του πληθυσμού, η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, οι σημαντικές διαφορές στο επίπεδο προστασίας της υγείας και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Θα πρέπει, παρά τα οικονομικά προβλήματα, να καταφέρουμε από κοινού να προσπαθήσουμε να ενιοποιήσουμε προς τα πάνω την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και θα πρέπει επίσης και τα συστήματα υγείας να έχουν συγκεκριμένο μέλλον και αυτές πρέπει να είναι νομίζω οι προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας στον τομέα της υγείας. Να σταθώ λίγο τώρα στις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες ε, στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αρκετές νομικές δραστηριότητες, νομοθετικές δραστηριότητες. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της Ισπανικής και της Βελγικής Προεδρίας έγιναν σημαντικά βήματα προόδου για την μεταχείριση και την αντιμετώπιση των ασθενών διαμεθοριακά. Επίσης υπήρξαν και κοινέ προσπάθειες στον τομέα νομοθετικές, στον τομέα των φαρμάκων, σχετικά με την οδηγία για τις μετακινήσεις των ασθενών η οδηγία αυτή νομίζω, η πρόταση οδηγίας μάλλον είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Οι προσανατολισμοί οι οποίοι δίδονται από την οδηγία αυτή θα δώσουν την δυνατότητα νομικής ασφάλειας και νομικών εγγυήσεων για όλους τους εμπλεκομένους. Να θυμίσω εδώ ότι η Ουγγαρία έχει υποστηρίξει και τη δεύτερη ανάγνωση της συγκεκριμένη πρότασης οδηγίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα, οι συμβιβαστικέ προτάσεις που έγιναν δεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτρέπουν στην Βελγική Προεδρία να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να εφαρμοστεί, να γίνει δεκτή πρώτα και να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη οδηγία. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων οδηγιών υπήρξαν σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της προστασίας γύρω από τα φάρμακα και τις φαρμακευτικές ουσίες. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο επέδειξε. Χάρη σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας καταλήξαμε σε συμβιβαστικές λύσεις γρήγορα. Είμαι πεπισμένο ότι λόγω ακριβώ των νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της προστασίας από τις φαρμακευτικές ουσίες θα μπορέσουμε να βρούμε σημαντικέ λύσεις σε προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τον πληθυσμό όπως ε, οι συνέπειες από τη χρήση φαρμάκων κτλ. Και οι παρενέργειες επίσης. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν τους ε, ε, χρήστες των φαρμάκων, τους ασθενείς. Επίσης ε, και σε σχέση με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα ελπίζουμε ότι να μπορέσουμε μέσω της νομικής πρωτοβουλίας που παίρνουμε τον Φεβρουάριο να την ολοκληρώσουμε. Οι προτάσεις αυτές ήταν βασικοί στόχοι θα έλεγα με τους οποίους ε, ασχοληθήκαμε τον τελευταίο καιρό. Ένα άλλο θέμα είναι η σωστή ενημέρωση των ασθενών. Είναι κάτι το οποίο ε, αντιμετωπίζουμε σαν θέμα, δεν έχει ορμάσει ακόμα η επεξεργασία του Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σας ε, διαβεβαιώ θα ληφθούν υπόψη. Πάντως σε αυτή τη φάση η Προεδρία περιμένει ε, μια νέα πρόταση από πλευράς, διορθωμένη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή τη στιγμή γίνει αυτό, τότε θα συγκληθεί η αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου. Θα θεωρούσαμε σωστό τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασθενών να είναι το κέντρο της αναθεώρησης της συγκεκριμένης πρότασης. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς από τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι σύγητες του. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι προτάσεις οι διορθωμένες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι στη διάθεσή μας το ταχύτερο δυνατόν και από αυτή τη στιγμή και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα σε βάθος. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τα φάρμακα, όχι μόνο στον τομέα των φαρμάκων, αλλά και γενικότερα στον τομέα της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στην υγεία. και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλους τους τομείς της υγείας. Η στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει την σημασία που έχει ο συγκεκριμένο τομέα. Καταρχά, αντιμετωπίζουμε το θέμα επί τη βάση των ευρωπαϊκών αξιών, αναγνωρίζουμε το σύνδεσμο ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την υγεία, τη συμπερίληψη της υγείας σαν σημαντικό παράγοντα σε διάφορους πολιτικούς τομείς, και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υγεία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν όλες αυτές οι αρχές αποτελούν μια σωστή βάση για την βελτίωση των και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα λοιπόν χρόνια οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε προβλήματα όπως η ασφάλεια των ασθενών, των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ιδέα για μια ζωή με υγεία και θα πρέπει επίσης και οι πολίτες της τρίτης ηλικίας να μπορούν να διάγουν τον βίο τους με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γενικά να είναι τα πράγματα πιο ελαστικά, να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η Ουγγρική Προεδρία θα βασιστεί στα αποτελέσματα της προηγούμενης και θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Για την ασφάλεια στον υγειονομικό τομέα θα θέλαμε να πούμε ότι τα παιδιά ιδιαίτερα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το θέμα των εμβολιασμών είναι σημαντικό. Θα κάνουμε διαβούλευση από αυτού γιατί είναι πρόβλημα σημαντικό. Υπάρχει και το θέμα της επιτήρησης, της προσοχής της κατάστασης της υγείας των παιδιών μεταναστών θα οργανώσουμε από αυτού στη Βουδαπέστη μια διάσκεψη και τα συμπεράσματά της κατά τις 3-4 Μαρτίου και τα συμπεράσματά της θα διαβιβαστούν στις υγειονομικές υπηρεσίες των χωρών μελών. Και με βάση τα συμπεράσματα αυτά θα δούμε τι δραστηριότητες πρέπει να αναλυφθούν, τι μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο και θα συζητηθούν όλα αυτά και από το Συμβούλιο. Η υγειονομική κατάσταση των πολιτών πρέπει να βελτιωθεί, ιδιαίτερα για τα παιδιά που πρέπει να έχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζονται για να έχουν τον υγιέστερο δυνατό τρόπο ζωής. Η Ουγγρική Προεδρία θα ήθελε να συνεχίσει το δρόμο των προηγούμενων, σας το είπα αυτό. Η ψυχική υγεία επίσης είναι το ίδιο σημαντική με την σωματική και το Ευρωπαϊκό Κόμμα Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και των νέων διότι υπάρχει και ένα θέμα ψυχικών ασθενειών στον τόπο εργασίας. Πέντε θεματικές διασκέψεις θα οργανωθούν για τις πτυχές αυτού του προβλήματος και τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα θα εμφαίνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τελευταία από αυτές τις διασκέψεις θα γίνει στη, και αυτή στις 3 Μαρτίου, στο Βερολίνο όμως. Και μετά θα αρχίσει η συζήτηση στο Συμβούλιο. Θεωρούμε επίσης σημαντικό οι ανισότητες μεταξύ χωρών μελών στον τομέα της υγείας να διευθετηθούν ώστε η σωστή και υγιεινή διατροφή να προωθηθεί να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία, να προωθηθεί η σωματική δραστηριότητα και να καταπολεμηθεί το κάπνισμα. Στις 31 Μαΐου του 2011 θα οργανώσουμε τη σχετική διάσκεψη. Επίσης θέλω να τονίσω ότι σε συνδυασμό με το Eurosef και με τη στήριξη της Κομισιόν στις 16 και 17 Ιουνίου θα οργανωθεί διάσκεψη εμπειροχνομόνων για την πρόληψη ατυχημάτων θα γίνει μια ανάλυση της κατάστασης και θα δούμε τι πρέπει να γίνει για το μέλλον. Εξάλλου υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων υγείας. Το βασικό θέμα του προγράμματός μας για την υγεία είναι το υγειονομικό διαβατήριο των πολιτών. Για τους δε απασχολούμενους στον τομέα υγείας επίσης υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που όμως δεν απαιτούν διαμεθοριακή συνεργασία όπως η περίθαλψη μεταναστών, το θέμα των, του εργατικού δυναμικού στην υγεία γιατί πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις εκεί, πρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημα μιας ποιοτική υγειονομικής περίθαλψης και να λάβουμε υπόψη μας και τα δικαιώματα των ασθενών. Η Ουγγρική Προεδρία θα τα θίξει όλα αυτά. Το σημαντικότερο είναι να γίνουν επενδύσεις στα μελλοντικά υγειονομικά συστήματα διότι οι προϋπολογισμοί σε όλες τις χώρες έχουν περικοπεί ενώ ο πληθυσμός συνεχώς γυράσκει και είναι όλο και ακριβότερη η περίθαλψη. Φυσικά οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι απλές δαπάνες, είναι σαν επένδυση για το μέλλον. και στο μελλοντικά θα μειώσει το κόστος. Πρέπει λοιπόν οι αποφάσεις που λαμβάνονται να εφαρμόζονται κιόλα και να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή τους. Να γίνει ένας πραγματικός διάλογος και να διευρύνουμε τις γνώσεις που έχουμε για το θέμα. Να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια και από τα διαρθρωτικά ταμεία για να βελτιωθούν τα συστήματα υγείας. Η Ουγγρική Προεδρία θα κάνει θα διατυπώσει προτάσεις ώστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να εφαρμοστούν και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα, βιώσιμο σύστημα υγείας με σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών. Η Ουγγρική Προεδρία έχει πολύ συγκεκριμένε φιλοδοξίες εδώ. Θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος για την ειδικευμένη εργασία στον τομέα της υγείας παραδείγματος χάρη κάτι που άρχισε η Βελγική Προεδρία στα συμπαράσματα της οποίας θα βασιστούμε για να ζητήσουμε επενδύσεις για την πρόσληψη περισσότερων ασχολούμενων με την υγεία. Επίσης πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα δράσης όσο το δυνατόν συντομότερα και να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί ότι είναι ζωτικό να δοθούν πραγματικές πληροφορίες και δεδομένα για την κατάσταση των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη. Και επίσης να πάψει επιτέλους η διαρροή εγκεφάλων των υγειονομικώς απασχολουμένων. Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες υγείας και οι εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντικό θέμα και για τη διαμεθοριακή συνεργασία. για να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. Θέλουμε λοιπόν στις 10 και 12 Μαΐου να οργανώσουμε μία διάσκεψη στη Βουδαπέστη για αυτό το θέμα. Κατά τις διάφορες αυτές διασκέψεις και εκδηλώσεις θα καλέσουμε εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας και ελπίζω να ανταποκριθείτε θα σας καλέσουμε και εσάς ώστε να υπάρχει στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες αυτές τις προτάσεις. Και τώρα θα απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε Βοντά για την παρουσίαση αυτή. Δικαίως είπατε ότι το θέμα της υγείας είναι πολύ σημαντικό για όλους για όλους λέω. Προηγουμένως είχαμε ψηφίσει για το θέμα των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και ανησυχεί ιδιαίτερα. Οι διαφορές αυτές από χώρα σε χώρα ως προς την πρόσβαση στην περίθαλψη Έχουν ζητήσει ήδη πολύ το λόγο, ο καθένας μόνο δύο λεπτά. Αρχίζω από τον Ριχάρδο Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Προεδρία σας. Αναφέρατε πολλά σχέδια και προτάσεις για τις υγειονομικές υπηρεσίες και για τη διαμεθοριακή επ' αυτού συνεργασία και εμείς συχνά συζητούμε τέτοια θέματα και θα θέλαμε και εμείς όπως και εσείς να εφαρμόζονται και όλα όσα συζητούνται. Η κυρία Γκροστέτ και ο κύριος Μπόβης ιδιαίτερα το προσέχουν αυτό. Πρέπει και στο Συμβούλιο να εφαρμόζονται όλα αυτά και να γίνονται οι απαραίτητες ε, διευθετήσεις των οδηγιών. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ μας ως προς την κοστολόγηση των διαφόρων προτάσεων ας πούμε να είναι φτηνότερη περίθαλψη για τους οικονομικούς ασθενέστερους. και τις οικονομικώς ασθενέστερες. Διότι πολλοί και πολλές μπορεί να ζητήσουν περισσότερη πρόσβαση διαμεθοριακώς εάν υπήρχε, εάν είχε υπάρξει ένα σύστημα κάρτας υγείας που να τους διευκόλυνε τα πράγματα. Για τους δε απασχολούμενους στον τομέα της υγείας Είναι γνωστό ότι υπάρχουν μεταναστευτικές ροές και άρα αυξημένη ζήτηση ιατρών και νοσοκόμων. Το θέμα της υγείας των παιδών επίσης είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερα για την πρόληψη, γιατί και αυτό είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η υγεία του πληθυσμού. Έγινε λόγος για ανισότητες των συστημάτων. Είδαμε τι έγινε με την επιδημία της γρήπης πέρυσι αλλά και φέτος και δεν νομίζετε ότι πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμός και φέτος μια καμπάνια εμβολιασμού. Δεύτερον, Υπάρχει η περίπτωση μίας μέας στην Ουγγαρία που συνελήφθη και κρατείται κατοίκον πριν από τα Χριστούγεννα μόλις και μετά μεταφέρθηκε σε μια φυλακή υψηλής ασφαλείας. Στην Ουγγαρία είναι νόμιμο να γίνονται γεννήσεις κατοίκων αλλά δεν υπάρχουν διατάξεις που να διέπουν το επάγγελμα της ΜΕΑΣ. Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτή η ΜΕΑ κατηγορείται και πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένα νομοσχέδιο, ένας νόμος που να επιτρέπει την κατοίκον γέννηση χωρίς να χρειάζονται τόσες πολλές άδειες Αυτά τα είπαμε και το Δεκέμβριο. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους διεθνώς. Εγώ έχω λάβει πολλά γράμματα και μηνύματα που μου λένε πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αντωνία Παρβάνοβα. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό για την παρουσίαση την οποία έκανα. Όταν έρχονται οι υπουργοί εδώ μας λένε καλά λόγια, αλλά η κατάσταση στον τομέα της υγείας δεν είναι καλή. Οι φιλοδοξίες πάντως της Προεδρίας είναι θα έλεγα κάτι το ιδιαίτερα θετικό και στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και στον τομέα της διαχείρισης της κρίσης την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουν τα συστήματα υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις οποίες θα πάρετε. Πώς θα συζητήσετε τον τομέα της υγείας στο Συμβούλιο, γιατί υπάρχει μία μόνιμη, θα έλεγα, διστακτική θέση του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Στην ουσία κρύβεστε εσείς εννοώ στο Συμβούλιο πίσω από την αρχή της επικουρικότητας. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εάν πράγματι θέλουμε να καλύψουμε την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό και αηφόρο σύστημα υγείας. Η Επιτροπή μας σήμερα το πρωί υιοθέτησε μια σημαντική γνωμοδότηση σχετικά με, τις, με τους τύπους της γρήπης που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και απαιτείται να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα από τις πανδημίες αυτές έτσι ώστε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω, μιας και η Επιτροπή επίσης ασχολείται με το θέμα, τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Σκοπεύετε να ενισχύσετε ε, τον σεβασμό των κανόνων διαφάνειας, και τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων σε περίπτωση που ξεσπάσει μια μείζον κρίση στον τομέα της υγείας. Σήμερα το πρωί εμείς ψηφίσαμε κατά ουσιαστικά της αρχής αυτής. Σκοπεύετε να το θέσετε σε συζήτηση έτσι ώστε για τους εμπειρογνώμονες αυτούς να γνωρίζουμε περισσότερα το παρελθόν τους όπως επίσης και τις προθέσεις τους. Κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω ε, είναι κάτι που αφορά και την, ε, το ζήτημα της ε, μετακίνησης της αρμοδιότητα, αρμοδιότητας για, τα γενετικά, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς α, στην, στον τομέα του Επιτρόπου Υγείας. θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εμείς έχουμε εκτιμήσει ότι αυτή η μετακίνηση ήταν ένα για να πάψει να έχει αρμοδιότητα ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ε, και να συνεχίσουμε τη στάση που είχε στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλές χώρες που όπως γνωρίζετε έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στην καλλιέργεια των γενετικά τροπομένων οργανισμών. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό απλώς ως ζήτημα υγείας των καταναλωτών ή και υγείας ε, των ε, οικοσυστημάτων και προστασίας της βιοπικιλότητας. Αν λοιπόν έχετε μια αντίστοιχη προσέγγιση ε, στη χώρα σας και πώς αυτό θα το εκφράσετε σε συγκεκριμένες πολιτικές παρακολουθώντας την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών που είναι αρνητικοί στα γενετικά τροποποιημένα τροποποιημένα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Sì, grazie, grazie Presidente. Allora, come lei saprà, abbiamo un γνωρίζετε ότι εμείς ψηφίσαμε ένα έγγραφο σήμερα σχετικά με το δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να πηγαίνει να θεραπευθεί σε οποιαδήποτε χώρα θέλει. Αν ένας πολίτης όμως πάει σε μια άλλη χώρα, τι ακριβώς συμβαίνει και όταν το κάνει αυτό μόνο και μόνο για να αποφύγει ας πούμε τους, ε, την ε, ουρά σε εισαγωγικά η οποία μπορεί να υπάρχει στη χώρα προέλευσης και το κόστος εδώ πώς θα καλυφθεί. Μπορεί να υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εδώ διαφορά ανάμεσα στο κόστος από τον ένα χώρο στον άλλο, από τη μία χώρα στην άλλη και την διαφορά αυτή καλείται να την καλύψει ο πολίτης. Όταν ένας πολίτης μπορεί λοιπόν να πάει σε μια άλλη χώρα θα το κάνει αυτό πληρώνοντας τη διαφορά του κόστου. Στην ουσία λοιπόν δεν δώσαμε μια πραγματική λύση σε αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας αλλά και οικονομικά προβλήματα. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό δεν είναι σωστό και δεν διασφαλίζει την ισότητα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζοντας βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στα κρατη και είτε να τροποποιηθεί η συνθήκη σχετικά με τις εθνικές αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας ή να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν εγγυημένες κατελάχιστον τουλάχιστον υπηρεσίες υγείας Κάποιες χώρες που έχουν περισσότερες δυνατότητες να πάνε πιο μπροστά, αλλά να υπάρξουν κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις για μια αρρωγή, θα έλεγα αντίστοιχη, ε, σε κάθε χώρα. Ποιες είναι οι απόψεις σας λοιπόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό σε κάποια ελάχιστα επίπεδα ευρωπαϊκής πρόνοιας στον τομέα της υγείας. Ο κύριος Ρέτελνη. Ο Υπουργός έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να, μιλήσω στο, να απαντήσω στον κύριο Ζέμπερ πρώτα. θέσατε μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι η Ουγγρική Προεδρία σκοπεύει να κάνει ό,τι περνάει από τις αρμοδιότητές της και από τις δυνατότητές της έτσι ώστε η οδηγία για τις μετακινήσεις των ασθενών να μπορέσει να γίνει δεκτή, να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αναφερθήκατε επίσης και στο θέμα της υγείας online και είπατε ότι είναι κάτι το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να διευκολύνει και το θέμα των μετακινήσεων των ασθενών πέραν των σύνορων. Έχετε δίκιο, θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στα πλαίσια μίας από τις συναντήσεις ε, που προβλέπουμε. Για τα θέματα της υγείας των παιδιών και για το θέμα της έλλειψης των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα υπάρχουν εδώ βαθύτατες ανισότητες. Ανισότητες τις οποίες θα πρέπει επιτέλους να προσπαθήσουμε να καλύψουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι εξηγεί την αναχώρηση, την αποχώρηση των ιατρών από μία χώρα και τη μετακίνησή τους σε μία άλλη χώρα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση αυτών των μεταναστευτικών τάσεων που επιδεικνύει το ιατρικό προσωπικό. Για να επανέλθω στα θέματα της υγείας των παιδιών, εμβολιασμοί και πρόληψη. Σε ορισμένες χώρες οι πολιτικές εμβολιασμού, σαν παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Υπάρχουν από την άλλη χώρες στις οποίες υπάρχουν σαφέστατα κενά οφείλουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις προϋποθέσεις της υγείας των παιδιών και της ασφάλειας της υγείας των παιδιών έτσι ώστε κάποιες ασθένειες οι οποίες μπορούν να καταπολεμηθούν μέσω του εμβολιασμού να είναι διαθέσιμες οι δράσεις αυτές και να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όπου αυτό, να εμβολιάσουμε όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Μακέβαν για τη γρήπη των χείρων, πρέπει να μελετήσουμε το ρόλο των διαφόρων φορέων, των διαφόρων οργανισμών και να καθορίσουμε ακριβώς το ρόλο τους. Όσον αφορά τώρα την ε, προμήθεια σε εμβόλια, πρέπει να το εξασφαλίσουμε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια άνηση κατάσταση όπου ορισμένα κράτη-μέλη θα έχουν πλεόνασμα και άλλα κράτη-μέλη έλλειμμα ή να έχουν εμβόλια τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Σχετικά με τις ΜΕΕΣ στην Ουγγαρία, υπάρχει ένας νόμος τώρα στην Ουγγαρία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς μια γυναίκα να γεννήσει στο σπίτι το και δηλαδή κατοίκων. Ο νόμος ε, αυτός ορίζει τις προϋποθέσεις, τους κανόνες και οι υπουργοί έχουν ήδη συζητήσει το νομοσχέδιο αυτό και τώρα θα πάει σύντομα στη Βουλή. Τώρα γιατί η κυρία Γκέρι βρίσκεται σε υποκράτηση ή στην φυλακή δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα όταν αντιμετωπίσαμε αυτή την περίπτωση οι αρμόδιες αρχές ενήργησαν πάρα πολύ γρήγορα και διαβουλεύτηκαν με οργανώσεις πολιτών, με ε, δημόσιες αρχές. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στην Ουγγαρία που είναι υπέρ του τοκετού στο σπίτι. Ε, ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις και ε, μετά από αυτό το διάλογο ε, δημιουργήθηκε αυτό το νομοσχέδιο, προτάθηκε αυτό το νομοσχέδιο που θα ρυθμίσει την όλη κατάσταση και ελπίζουμε να περάσει. Η κυρία Αντώνια Παρανόβα. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα των Υπουργών Υγείας να το ακούσουν οι Υπουργοί Οικονομικών. Στην συνεδρίαση ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου τέθηκε αυτό το ζήτημα και επίσης συζητήσαμε το ενδεχόμενο το ΕΚΟΦΗΝ και η ΕΠΣΚΟ να κάνουν μια κοινή συνεδρίαση. Το μήνυμα των Υπουργών Υγείας για τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι θα πρέπει οπωσδήποτε τα θέματα υγείας να καλυφθούν από το πλαίσιο αποφάσεων, των οικονομικών αποφάσεων για τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά εθνικά θέματα. Για να ξεπεραστεί η κρίση χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση του τομέα της υγείας. ο τομέας της υγείας είναι ένα απίστευτα περίπλοκο θέμα, πρέπει να το γνωρίζουμε σε βάθος, να ξέρουμε όλες τις πτυχές των ε, απασχολούμενων στον τομέα της υγείας, των αρρώστων, των ε, υγειονομικών φορέων. Όταν ξέρουμε λοιπόν σε βάθος όλους, όλες τις πτυχές θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ενδεχομένως τις κρίσεις στο μέλλον. Όσον αφορά το ΙΤΑ 1, 1, τη γρήπη των χείρων, ε, πρέπει να, να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες των ε, τελευταίων ετών, τις πρόσφατες εμπειρίες. Ο κύριος Τέμπαλος έστειλε, ε, έθεσε ένα θέμα για τα γενετικά τροποποιημένα. Είναι και αυτό ένα περίπλοκο ζήτημα. Πρόκειται για την αγροτική οικονομία, την υγεία του περιβάλλον και ε, πρέπει να τονίσουμε το, την πτυχή της υγείας. Τη διάσταση της υγείας. Δεν θα θέσουμε το θέμα αυτό ξεχωριστά στην ημερήσια διάταξη της Ουγγρικής Προεδρίας των επόμενων έξι μηνών τα γενετικά τοποποιημένα, αλλά θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο της υγείας. Ε, το τελευταίο ερώτημα αφορούσε ε, τον ελάχιστο τα, τα ελάχιστα πρότυπα στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα ζητήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα ελάχιστα standards. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές λοιπόν μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να προσέξουμε εμείς ιδιαίτερα να αμβλύνουμε αυτές τις μεγάλες διαφορές, να μειώσουμε αυτές τις μεγάλες διαφορές στα κράτη όπου οι βασικές υπηρεσίες δεν είναι τόσο αναπτυγμένες. Ε, εκεί πρέπει να σηκώσουμε, να ανεβάσουμε το επίπεδο των βασικών υπηρεσιών, να τις βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε επίσης και τα προσόντα του προσωπικού υγείας αυτές οι ανισορροπίες στον τομέα της υγείας πρέπει να επισημανθούν, πρέπει να αναλυθούν και να δημιουργηθεί ένας κατάλογος προτεραιοτήτων εξάλληψης αυτών των ανισοτήτων. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μία κρίση που αφορά όλες τις πτυχές της κοινωνίας και πρέπει να εξασφαλίσουμε η κρίση αυτή να ζημιώσει τον τομέα της υγείας όσο το δυνατόν λιγότερο Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο για τι απαντήσει. Ο ε, δεύτερος γύρος, ο Μύροσλαβ Νικολάσικ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, ε, απευθύνεσαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει και προβλήματα, τα θέματα της υγείας και της κρίσης, τους μεγάλους κινδύνους στον τομέα της υγείας. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία. Είμαι πολύ ευτυχής που αναφέρετε τα τα ταμεία και τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά μέσα. Και τη δυνατότητα να ε, ε, αναλύσουμε λίγο περισσότερο τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση για όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης αναφέρατε την πρόληψη σε σχέση βεβαίως με τον τρόπο ζωής, με το lifestyle και αναφέρατε και τη νέα γενιά, τη νεότερη γενιά. Η Φιλανδία και η Ουγγαρία δυστυχώς είχαν έναν υψηλό αριθμό αυτοκτονιών μεταξύ του νέου πληθυσμού. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν έχετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Και το συγκεκριμένο μου ερώτημα για αυτή τη συνεδρίαση είναι ποιες είναι οι απόψεις της Ουγγρικής Προεδρίας για το αυξανόμενο μεταναστευτικό κύμα ε, η προσωπικού υγείας και επιστημόνων ε, που φεύγουν από την Ουγγαρία για άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρουοτ Μπέρεντ. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσουμε το θέμα του μεταναστευτικού κύματο στον τομέα της υγείας. Πρέπει να ξέρουμε γιατί γίνεται, γιατί σημειώνεται αυτό το κύμα μετανάστευση. Είμαι πολύ περίεργη να γνωρίσω τους λόγους. Μήπως ξέρετε εσεί, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, πέρα δηλαδή της, των χαμηλών εισοδημάτων και της δυσκολίας ε, απασχόλησης, δεν ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το ρεύμα μετανάστευσης. Επίσης θα ήθελα να πω ότι τα προγράμματα που, που παρουσιάσετε είναι σωστά, δεν είναι υπερβολικά φιλόδοξα για έξι μήνες, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά ε, θα ήθελα να ξέρω εάν, ε, εάν πιστεύετε πραγματικά ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα του e-health, δηλαδή της ε, ηλεκτρονικής υγείας ε, και της διασυνοριακής, των διασυνοριακών υπηρεσιών. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα γιατί το Συμβούλιο μας ε, μπλοκάρισε διασυνοριακές παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας. Και κάτι για την ομοθεσία, αυτό θα το για τα γενετικά τοποποιημένα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Βάζεκας αύριο ε, ελπίζω να συνεχίσετε με ορμή το νομοθετικό πρόγραμμα, αλλά έχω λίγο απογοητευτεί για το θέμα των ασθενών. Είπατε ότι πρέπει να περιμένετε την τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν θα σας πει ήδη τι θα περιλαμβάνει η πρότασή της που προσεγγίζει την άποψη του Κοινοβουλίου. Ήδη χάσατε τέσσερις εβδομάδες και ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και μας καίει ιδιαίτερα είναι τα συμφέροντα των ασθενών και η προάσπιση των ασθενών. Γι' αυτό θα ήθελα το ταχύτερο να συγκαλέσετε την ομάδα εργασίας διότι αν η Κομισιόν έρθει σε εμά με την τροποποιημένη πρόταση και αρχίσετε την εργασία το Μάρτιο, μέχρι το τέλο τη Προεδρία δεν θα μπορέσετε να καταφέρετε τίποτα και αυτό θα είναι πολύ λυπηρό. Ο πρόεδρο, η κυρία Λεπάζου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Με έκπληξη είδα ότι δεν έχετε στο πρόγραμμά σας τα γενετικώς τροποποιημένα. Αν και σε οδηγία του 2008 συζητήθηκε το πράγμα, ξέρω ότι είναι λεπτό πρόβλημα, αλλά με εκπλήσει ότι δεν συζητιέται καν στην Προεδρία σας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που θέλω να συζητήσω εδώ. Θέλω να πω περίπου αυτά που είπε η κυρία Παρβάνοβα. Η διαχείριση της κρίσης, μάλιστα μια τόσο σημαντική όσο αυτή με το φάρμακο Μεντιατόρ στη Γαλλία, η χρήση των φαρμάκων, είναι κάτι που πρέπει επίσης να χειριστούμε. Το πρωί δεχτήκαμε μια έκθεση που ζητά υποχρεωτική δημοσίευση των συμπερασμάτων ειδικών για τέτοια προβλήματα πριν από δύο εβδομάδες στο Κοινοβούλιο μας είπε ένας εμπειρογνώμων ότι ένας επίτροπος ότι μπορεί να ζητήσει να ληφθούν υπόψη ε, τα συμφέροντα που δεν έχουν δηλωθεί και από την Γαλλική Υπηρεσία ΕΦΣΑ και αλλού. Γιατί αυτό που υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματός μας είναι ακριβώς αυτό και την, και την εμπιστοσύνη του πληθυσμού. Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα κύριε Υπουργέ να σας ζητήσω το εξής. Ε, η Προεδρία έχει σκοπό να σας ρωτήσω το εξής. Έχει σκοπό να κάνει τίποτε για αυτό το θέμα της ασφάλειας των φαρμάκων με συγκεκριμένες προτάσεις. Ε? Νάσα Τσίλντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Και εμένα με ενδιαφέρει η ψυχική υγεία. Το Μάρτιο είπατε ότι θα διοργανωθεί η σχετική διάσκεψη. Η Ουγγρική Προεδρία τι θα κάνει ώστε να διασφαλίσει ότι η συνεργασία μεταξύ ενδιαφερομένων και χωρών μελών, πράγμα που ζήτησε το Κοινοβούλιο επανειλημμένως, θα εφαρμοστεί και θα συνεχιστεί και θα ενδυναμωθεί θα ενθαρρύνει την Κομισιόν να κάνει τη σχετική πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Πιτέλα. Όχι. Ο κύριος λέει μάλλον. Κύριε Πρόεδρε, το, το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας είναι αρκετά φιλόδοξο. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνεργασία με την ομάδα εργασίας καταπολέμησης του καρκίνου. Δεν πρέπει όμως να μιλάμε μόνο για ασθενείς αλλά γενικότερα για πολίτες. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και οι υγιείς μπορεί να κινδυνεύουν. Μόνο έτσι θα μειωθεί ο αριθμός των ασθενών αν λάβουμε υπόψη μας και τους υγιείς. Χρειάζεται λοιπόν να συνεχιστεί η εργασία της μιας Προεδρίας από την άλλη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομίσκα. Χαιρετίζω την πρόθεσή σας να συμπληρωθεί η διαδικασία για την οδηγία, για την υγεία ως το δυνατόν συντομότερα. Αυτό είναι τελείως απαραίτητο και για τους ασθενείς και γιατί υπάρχει η αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται από μία χώρα στην άλλη. Μόνο αν υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα και της γνώσης θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλύτερη περίθαλψη. Σας ερωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ. Ποιο θα είναι το μεγαλύτερο όφελος των μέτρων σας. Ωραία ο Ζιλ Πανιό ακόμα στο δεύτερο γύρο και μετά θα δώσω το λόγο στον Υπουργό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα σήμερα το πρωί μία παρουσίαση γεμάτη καλές προθέσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να τονίσω ότι υπάρχει και αρκετά μεγάλη δυσθυμία εδώ, γιατί Γνωρίζουμε ότι στον τομέα της υγείας, στα πλαίσια αυτής της αρχής του 21ου αιώνα, πολλά είναι τα προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε την γρήπη πέρυσι ήταν ένα σκάνδαλο. Το φάρμακο Mediator στην Γαλλία είναι και αυτό ένα σοβαρό σκάνδαλο και τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι εμφανίζεται ένα νέο σκάνδαλο με την ουσία ασπαρτάμι που φαίνεται ότι η σημερινή κατανάλωση, η καθημερινή συγγνώμη κατανάλωσή του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Από την επικαιρότητα αυτή λοιπόν πρέπει να υποφεληθεί η Ουγγρική Προεδρία έτσι ώστε να πάρουμε τα πολιτικά μέτρα που θα επιτρέψουν να νιώσει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι προστατεύεται γιατί έχει την αίσθηση ότι είναι εκτεθειμένος. Διερωτώμε λοιπόν τι συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνεται σε επίπεδο ε, νομοθετικό έτσι ώστε να καλύψετε τις ανάγκες, τι περαιτέρω μορφές συντονισμού μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στα προβλήματα τα οποία όλοι αντιμετωπίζουμε σήμερα ελπίζοντας έτσι να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να καταλήξουμε στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν σε πολλές ε, χώρες. Εκπλήσωμαι επίσης και από την απάντηση που δώσατε για την ε, ε, ΜΕΑ στην Ουγγαρία. Εσείς σας θυμίζω έχετε καταδικαστεί από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τέτοιου ίδιους ρυθμίσεις. Και γιατί δείξατε μια τέτοια άγνοια του θέματος. στην απάντησή σας δεν το κατανοώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καταρχά τον κύριο Νίκολα απαντώ. Θα ήθελα λοιπόν να πω στο θέμα της πρόληψης και υγιούς ε, τρόπου ζωής. Το συνέδριο το οποίο θα οργανώσουμε για αυτά τα δύο θέματα, πρόληψη και lifestyle, ε, αφορά τους πολίτες, ε, την υγεία των πολιτών και δι των νέων, πιο νέων, της νέας γενιάς. Διότι αυτά τα δύο πάνε μαζί, η πρόληψη και ο τρόπος ζωής στους νέους και θα συμπεριλάβει και την ε, ψυχική υγεία. αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την ψυχική υγεία και, την, ε, και, τον καλό τρόπο ζωής ε, συμφώνησα και στο συνέδριο αυτό που θα διοργανώσουμε θα ασχοληθούμε ακριβώς με όλες τις πτυχές της ευζωίας, της ψυχικής υγείας και του τρόπου ζωής. Ε, αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και πιστεύω πιστεύουμε ότι πρέπει η νέα γενιά να προετοιμαστεί κατάλληλα μέσω της παιδείας ώστε να έχει μία ψυχική στήριξη ε, στο θέμα των ε, αυτοκτονιών ακριβώς που ρωτήσατε πρέπει καταρχάς να εντοπίσουμε τα αίτια και συνεχεία να δουλέψουμε πάνω στην πρόληψη. Η μετανάστευση, το μεταναστευτικό κύμα, απαντώ σε όσους ερώτησαν, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός. Ε, βεβαίως έχει σχέση το, η μετανάστευση αυτή και με την αγορά εργασίας και με το επίπεδο εισοδημάτων. Ε, πρέπει να ενισχύσουμε τον τομέα της υγείας. Ε, πώς μπορούμε να, να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε την ειδίκευση των γιατρών, του ιατρικού προσωπικού, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή τους, ε, την, ε, τις ειδικότητε, να διευρύνουμε τις ειδικότητε. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια στατιστικών αναλύσεων ε, του φαινομένου αυτού για να καταλάβουμε γιατί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό φεύγουν από τη χώρα. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις απόψεις τους και να καταλάβουμε τα αίτια, το, τους λόγους για τους οποίους φεύγουν. Η, το μεταναστευτικό κύμα είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτούς τους τομείς ε, ε, νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών από Ανατολή προς Δύση, ε, από Ευρωπαϊκή Ανατολή προς Ευρωπαϊκή Δύση νομίζω ότι μόνο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των ειδικοτήτων και τη βελτίωση της οικονομίας μπορούμε να ανακόψουμε αυτό το κύμα. Έχουμε πρόθεση να διοργανώσουμε ένα συνέδριο για αυτό το θέμα ε, επίσης. Τώρα, για το e-health, e-health ε, ηλεκτρονική υγεία. Ναι. Ε, μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες και διασυνοριακά να γίνει μια σωστή χρήση των ε, ε, διασυνοριακών συστημάτων υγείας, πληροφόρησης, ενημέρωσης των ασθενών από άλλες πηγές και γι' αυτό θα προσέξουμε και αυτό το θέμα, το e-health. E-health, ε a, a, a, a GMO-k, Lepázs asszonynak válaszolva, a... Η, η κυρία Όσον αφορά τους ε, γάμα μη όμικρον, αυτό αφορά την υγεία των πολιτών και θα συνεργαστούμε στενά με τους συναδέλφους, ε, τους αρμόδιους συναδέλφους, τους μάλλον συναρμόδιους. Για τη γρήπη των χείρων ε, πρέπει να ενισχύσουμε τα, τους ευρωπαϊκούς φορείς για την αντιμετώπιση. Το έχουμε υπόψη μας. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να έχει εμπιστοσύνη το κοινό, το, οι πολίτες μας, εμάς η κυρία Children's ε, έθεσε ένα ερώτημα για την ψυχική υγεία. Ε, είναι και αυτό προτεραιότητα. Ναι, ναι, όχι, είναι το πιο απλό. Και θα προ... διατυπώσουμε συμπεράσματα του στο Συμβούλιο όσον αφορά τον αντικαρκυνικό αγώνα Ε, πρέπει να βελτιωθεί και ο τομέας της υγείας και η, να αυξηθούν ε, τα κονδύλια, ε, οι πιστώσεις για τον τομέα αυτών. Η Βελγική Προεδρία υιοθέτησε συμπεράσματα στο Συμβούλιο και στα συμπεράσματα αυτά συμφώνησε η Ουγγαρία και βάσει αυτών των συμπερασμάτων ναι. θα εργαστούμε στον κοινό αντικαρκυνικό αγώνα. Υπάρχουν εθνικές αντικαρκυνικές εκστρατείες και αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θέλουμε να τονίσουμε την πρόληψη ιδιαίτερα και ε, τους συστηματικούς ελέγχους υγείας, τα check-ups των πολιτών. Ο κύριος Μπάνιο ανέφερε τα σκάνδαλα και πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε την επανάληψη σκανδάλων. Δυστυχώς αυτά τα σκάνδαλα αφορούν πολλούς πολίτες είναι σήματα αυτών των σκανδάλων και πολλοί κόσμος ανησυχεί για αυτή την κατάσταση. Το Συμβούλιο πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποφύγει αυτά τα προβλήματα, τα οποία οδηγούν σε μεγάλα σκάνδαλα. Όσον αφορά τη γρήπη, ναι. Ναι. Ήδη είπα, έχω ήδη αναφέρει ότι έχει αρχίσει η αξιολόγηση του, του φαινομένου και πιστεύουμε ότι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση της Ουγγαρέζας ΜΕΑΣ, ε, δεν μπορώ τώρα να απαντήσω εγώ εκ μέρους των Ουγγρικών Αρμοδίων Αρχών. Για αυτή την περίπτωση υπήρχαν όμως ε, στοιχεία στην περίπτωση αυτή που έδειξαν ότι η ΜΕΑ αυτή δεν ενήργησε σωστά και γι' αυτό ακριβώς ε, ε, οι αρμόδιες αρχές αντέδρασαν όπως αντέδρασαν. Σας είπα ότι όταν ε, ήρθαμε όταν ε, βρεθήκαμε εν γνώση αυτής της ε, περίπτωσης, αρχίσαμε αμέσως το διάλογο, διατυπώσαμε αυτό το νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να αγγιθούμε την ασφάλεια των γυναικών που επισημούν να γεννήσουν στο σπίτι τους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο ασφάλειας και για τη γυναίκα και για τον νεογέννητο. Ο πρόεδρος. Έχουμε αναλάβει πολλές πληροφορίες σε αυτό το θέμα του ε, τοκετού ε, κατοίκων. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ε, ερευνηθεί το θέμα αυτό περισσότερο σε βάθος. Χρειαζόμαστε ακόμα 40 υπογραφές για να περάσει αυτή η πρότασή μας από την Ολομέλεια. Πάντως έχουμε ασχοληθεί και δεσμευτεί πολύ σημαντικά. 27 χώρες ε, πιστεύω ότι πρέπει να συγκεράσουν τις προσπάθειές τους για να καταλήξουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Ο ε, τελευταίος γύρος ερωτήσεων, ο συμπατριώτης σας, ε, Γιάννος Έντερ. ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να θέσουμε του τρίτου γύρου. Δύο ερωτήματα έχω. Κύριε Υπουργέ, στην εισαγωγική σας ομιλία είπατε ότι υπάρχουν αυτές οι μεγάλες ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, πολλοί άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα. Εγώ ήθελα απλώς να συμπληρώσω και να πω εάν διαβλέπετε μία δυνατότητα να βοηθήσουν τα διαθροτικά ταμεία στην άμβληση αυτών των ανισοτήτων. Δεύτερη ερώτηση και πάλι στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε και άλλοι μίλησαν για το πόσο σημαντικός είναι ένας υγιής τρόπος ζωής ε, και για τους Ούγγρους πολίτες και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπατε ότι τι θέλετε, τι, τι προτίθεστε να πράξετε ένα τμήμα των πρωτοβουλειών σας, ένα μέρος των πρωτοβουλειών σας είναι η αντικαπνιστική εκστρατεία. Είμαι ε, τεταγμένος υπέρ του αντικαπνιστικού αγώνα και πολλοί άλλοι συνάδελφοι είναι. Θα ήθελα να ξέρω συγκεκριμένα τι έχετε πρόθεση να πράξετε κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Ιδίως για τη, τους νέους, δεδομένου ότι το κάπνισμα κερδίζει έδαφος στη νέα γενιά. Ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρο, ήσασταν πολύ σαφή και σύντομο. Ε, κύριε Υπουργέ, λέει ο κύριο Σνέλχαρτ, ε, <laughs> θα ήθελα να συνεχίσω με το θέμα των διαφορετικών ταμείων. Και εμένα με ενδιαφέρει πολύ η συμβολή τους. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω πού ακριβώς θέλετε να παρέμβει ε, το, τα διασωτικά ταμεία να παρέμβουν. Είναι για την διοργάνωση των ε, συνεδρίων, των διασκέψεων ή θέλετε, ε, μιλάτε για κονδύλια, για πιστώσεις οι οποίες θα διατεθούν στις υποδομές. Μιλήσατε για την υγεία των παιδιών και την παροχή υπηρεσιών για τα παιδιά, εμβόλια είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζονται τα κράτη-μέλη πολύ διαφορετικά. Ε, θέλετε να κάνετε τη συζήτηση αυτή ε, και να τη βάλετε στην ατζέντα του Συμβουλίου. Αυτή τη, το συνέδριο που αποφασίσατε να κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε όμως να επιβάλλουμε όλες, να, εφαρμόσουμε όλες αυτές τις προφορίες που έχουμε μαζέψει στην Ευρώπη και τελευταία ερώτηση όσον αφορά ασθενείς και επαγγέλματα στην Ευρώπη. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό το θέμα, ασθενείς και ε, επαγγελματικός ιστός. Η κυρία Κλάς, κύριε ε, Πρόεδρε του Συμβουλίου. Έχετε παρουσιάσει εδώ μία μεγάλη βεντάλια θεμάτων ε, και βλέπετε ότι αυτά που μας ενδιαφέρουν συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές. Ε, τρόπος ε, ζωής, ε, χρησιμοποίηση, δραστηριοποίηση των διαθροτικών ταμείων, εμβόλια, παροχές πλησιών στα παιδιά, για παιδιά, Όλα αυτά τα θέματα άπτονται του υγιού τρόπου ζωής με τη βοήθεια του, του πλαισίου υγείας. Αν ο νους ε, υγιής εν σώματι υγιή όπως λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Και ε, θα ήθελα να ξέρω πώς θα συνδυάσετε όλα αυτά τα θέματα. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι καθαρά πρόβλημα του τομέα της υγείας, αλλά είναι ένα καινούριο φαινόμενο και πρέπει να το συμπεριλάβουμε στα θέματά μας. Η περαιτέρω ανάπτυξη των διαφορετικών ταμείων είναι λίγο ασαφές αυτό το θέμα. Ενδιαφέρουσα η πρόταση, αλλά πιστεύω ότι πολλά ήδη έχει κάνει το Συμβούλιο, πολλές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Ε, έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως με τους αγροτικούς γιατρούς, με την έξοδο από τις, με την εσωτερική μετανάστευση από αγροτικές περιοχές. Και έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί δεν υπάρχει ε, σε όλη την Ευρώπη ένα σωστό σύστημα κροτικών ιατρίων όπου ο γιατρός μπορεί να κάνει και τις επισκέψεις στο σπίτι των ασθενών κλπ. Μήπως θα μπορούσε λοιπόν αυτό το θέμα να το αναπτύξετε. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε, αλλά πρέπει να βρούμε νέους και νετονικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ευχαριστώ. Δεν λέω, έχουμε αναπτύξει πολλές πρωτοβουλίες μεταξύ των οποίων όμως ο αγροτικός ιατρός, ο ιατρός του χωρίου όπως λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικός, αναφυσβήτητα. Ο κύριος Φλόρενς. Ε, πολλές φορές εδώ έχουμε υποστηρίξει αντικαρκυνικούς αγώνες, αλλά αντικαρκυνικές εκστρατείες. Δεν ξέρω ε, όμως, εάν Ποια είναι τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι αναφερθήκατε ότι θα τους περιλάβετε στο φάκελό σας. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα σε, μια, σε ένα κράτος μέλος, όπως η Γερμανία αυτή τη στιγμή υπάρχει το ποινικό αδίκημα των, διοξινών, το οποίο θα πρέπει να τακτοποιήσει, να ξεκαθαρίσει δηλαδή το κράτος η σχέση μεταξύ του σκανδάλου των διοξινών και του γεγονότος ε, ότι ε, χίλιοι άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρώπη κάθε μέρα από καρκίνο των πνευμών, λόγω του καπνίσματος δηλαδή, για μένα είναι τεράστια η διαφορά αυτή. Ε, από τη μία πλευρά έχουμε ενδείξεις, από την άλλη έχουμε αποδείξεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς θα ε, χειριστείτε αυτό το θέμα το οποίο είναι τεράστιας ευθύνης ποια θα είναι η στρατηγική σας συγκεκριμένη, δηλαδή στον ε, αγώνα. Ευχαριστώ κυρία Ροντ Μπέρεντ. Το μόνο που θέλω να πω είναι να, αν μπορεί να απαντήσει ο, υπουργό, ο Υπουργός σε μένα για την ενημέρωση των ασθενών. Δεν θα έπρεπε να είχατε αρχίσει ήδη άτυπα την ε, εργασία με την Κομισιόν για να μην καθυστερήσετε και παρουσιαστεί ένα αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας με την Κομισιόν το Μάρτιο για την ενημέρωση των πολιτών είναι το θέμα. Διότι μετά δεν προλάβατε τίποτα. Θα, θα, έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε, ήδη πρέπει να είχατε ξεκινήσει, να ξεκινήσετε την ομάδα εργασίας για την ενημέρωση των πολιτών αμέσως με την ε, Κομισιόν για να έχουμε αποτελέσματα. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Για να ακούσουμε και τις απαντήσεις τώρα. Σχετικά με το ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Γιάννος Άντερ και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των διαφθορτικών ταμείων είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών βουλευτών. Το θέμα δεν είναι να υπάρξει μια απλή οικονομική συνδρομή για την οργάνωση συγκεκριμένων συναντήσεων. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, των εξοπλισμών, των νοσοκομιακών για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Τους επόμενους έξι μήνες λοιπόν εμείς έχουμε θέσει σαν στόχο ακριβώς να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις διαφορές. Είναι μια προτεραιότητα αυτή για μας. Σχετικά με έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και ζωής. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την ε, διάδοση ακριβώς τέτοιων μορφών ζωής όπως επίσης ε, και την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων θυμίζω ότι υπάρχουν τρία θέματα εδώ, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στις συναντήσεις τις οποίες προανέφερα. Πρώτον, η σωστή διατροφή. Αυτό έχει άμεση σχέση με τον τρόπο ζωής φυσικά. Ένα δεύτερο είναι η γυμναστική και ο αθλητισμός. Και οι σωματικές δραστηριότητες, κάτι το πολύ σημαντικό όχι μόνο για τους νέους και τα παιδιά, αλλά και για την τρίτη ηλικία και οι πολίτες τρίτης ηλικίας θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ένα επίπεδο σωματικών ικανοτήτων ε, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και τρίτο θέμα είναι η κατανάλωση προϊόντων καπνού, το κάπνισμα. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να επηρεάσουμε τους νέους και να εμποδίσουμε την κατανάλωση ε, καπνού η οποία επεκτείνεται. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους, να τους δείξουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι των οποίων διατρέχουν για την υγεία τους. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από μέτρα λοιπόν, τα οποία έχουν σαν στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ε, προϊόντων ε, καπνού, ιδιαίτερα στους νέους, σαν παράδειγμα απαγόρευση καπνίσματος σε ορισμένους χώρους ή ε, περιορισμένη δυνατότητα σε χώρους, σε συγκεκριμένους χώρους κτλ. Τώρα για τον κύριο Σνέλχαρτ, ο οποίος έφτιασε ένα ερώτημα για τα διαφορετικά ταμεία, θα ήθελα συμπληρωματικά να πω ότι πράγματι έχουμε ανάγκη από περισσότερες επενδύσεις και για τους εμβολιασμού. Δεν μπορούμε εμείς να καταστήσουμε υποχρεωτικούς τους εμβολιασμού σε όλες τις χώρες, αλλά μπορούμε να τεκμηριώσουμε σωστά τα ωφέλη και τα θετικά των εμβολιασμών. Κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση και με την μετανάστευση και τα πιθανά μεταναστευτικά ρεύματα όπου θα πρέπει να υπάρχουν ε, βιβλιάρια εμβολιασμού πολύ πιο οργανωμένα από ό,τι σήμερα. Το θέμα των μεταναστευτικών ροών είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και σε σχέση ε, με, με το ιατρικό προσωπικό και το ε, νοσηλευτικό προσωπικό που θα πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν τα ειδικά προβλήματα αυτών των μεταναστευτικών ροών. ο γιατρός, ιδιαίτερα ο οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος αν θέλετε, θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα μέσα στην διάθεσή του και να μπορέσει να λειτουργεί ο παθολόγος με ποιοτικό τρόπο και να ωφελήσει έτσι το σύνολο του συστήματος υγείας. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την βελτίωση της ποιότητας μέσω της σωστής κατάρτισης του προσωπικού υγείας. Τα επαγγέλματα γύρω από τον τομέα της υγείας ε, είναι οργανωμένα με πολύ ιεραρχικό τρόπο Από τη μία ο ασθενής, από την άλλη οι ιατροί, οι νοσοκόμοι και το υπόλοιπο ειδικευμένο προσωπικό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τις ισορροπίες που υπάρχουν και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Οι μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού από τη μία χώρα στην άλλη είναι κάτι που πρέπει να μας αποσχολήσει λοιπόν και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Η Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσει να προτείνει κάποιες ε, σκέψεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Για την κυρία Κλάις. έθεσε και αυτή το θέμα των διαφθορτικών πόρων, των διαφθορτικών ταμείων. Είναι κάτι φαίνεται το οποίο απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάθος. Θα μπορούσε εδώ να απαντήσει κανείς λέγοντας ότι το θέμα ε, έχει πάρα πολύ, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλες τις ηλικίες και τους νέους και την τρίτη ηλικία συμπεριλαμβανομένων. Έχουν πράγματι υπάρξει δημογραφικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια που επηρεάζουν τον τομέα της υγείας με διάφορους τρόπους. Το πρόβλημα της δημογραφικής εξέλιξης της Ευρώπης τίθεται και γι' αυτό καλούμεθα να βελτιώσουμε την κάλυψη των αναγκών στον τομέα της υγείας των ε, πολιτών τρίτης ηλικίας, των ηλικιωμένων. Απαιτείται σωστή ενημέρωση, η οποία θα πρέπει να καλύψει όλους τους ενδιαφερομένους και η οποία θα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο. Θα πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος ζωής, ο σωστός τρόπος διατροφής, να γνωρίζουν τα παιδιά ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού τους και πώς μπορούν να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σώματός τους. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά, ε, τα οποία όταν γίνουν ενήλικοι θα γνωρίζουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος ζωής. Ε, για το κάπνισμα ήδη αναφέρθηκα σας είπα για το πρόγραμμα δράσης και για την ε, συνάντηση την οποία θα οργανώσουμε τη διάσκεψη γύρω από το θέμα ε, του καπνού. Σχετικά τώρα με το θέμα της ενημέρωσης των ασθενών, σας ευχαριστώ που μου θυμήσατε για δεύτερη φορά το συγκεκριμένο θέμα. Το είχαμε ήδη συζητήσει το Δεκέμβριο στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ουγγρικής Προεδρίας συνεργαστήκαμε με τον αρμόδιο επίτροπο και του ζητήσαμε να μας μεταφέρει τον φάκελο και όλα τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσουμε τις καθυστερήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που μας αναφέρατε το πρόγραμμά σας. Είδατε πόσο Δεσμευμένοι είμαστε έναντι της ε, προστασίας και της ασφάλειας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Η ενημέρωση των πολιτών είναι η μόνη νομοθετική πτυχή, το μόνο νομοθετικό ζήτημα το οποίο πιστεύουμε να, ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το εξάμεινο διότι είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση. Ε, κατά τα άλλα το πρόγραμμά μας είναι ευρύ αλλά ιδιαίτερα θα προσέξουμε και τις, την πρόληψη ε, που καλύπτει ε, τη σωστή διατροφή, σωστό τρόπο ζωής, όχι υπερβολική κατανάλωση, είναι ο πνεύματος και τονίσατε, τονίστηκε επίσης ε, η οξία ανισότητα ε, στον τομέα της υγείας, στους τομείς της υγείας των κρατών μελών, οι ανισότητες που υπάρχουν στην υγεία ε, και επίσης βεβαίως το μεταναστευτικό κύμα από τη χώρα σας και τα διαφορετικά ταμεία αναφέρθηκαν πολλές φορές. Σας ευχόμαστε καρποφόρο εργασία, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας αυτό το εξάμενο και ε, πιστεύουμε ότι πολλοί συνάδελφοί μας θα ενδιαφερθούν και θα συμμετάσχουν σε, αυτές τις ειδικές, σε αυτά τα ειδικά συνέδρια και ημερίδες που θα διοργανώσετε. Σας ευχαριστώ ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, ευρωβουλευτές, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να μπορέσουμε σύντομα να απαντήσουμε και στα ερωτήματα που δεν, μπορώ, δεν μπόρεσα σήμερα να απαντήσω 100%. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι θα είστε ικανοποιημένοι με την εξάμενη προεδρία μας. Θα συνεργαστούμε πολύ στενά μαζί σας και η καλή συνεργασία είναι η βάση ε, των καλών μας σχέσεων. Ευχαριστώ.